Well, thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ούτε τα παιδιά μου δεν με ακούνε τόσο καλά. Υπέροχα. Θα ήθελα λοιπόν να ανακοινώσω την έναρξη της συνεδρίασης και ελπίζω να μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρίς τροποποιήσεις. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχω αρκετές. Διατίθεται διερμηνία σε όλες τις γλώσσες ε, της Επιτροπής ε, Ήτρα και Ένβη, εκτός από κροατικά. Δουλέψαμε πολύ. Λάβαμε 920 τροπολογίες και έχουμε ένα φάκελο που ξεπερνά τις 500 σελίδες και για οικονομία χαρτιού όλη η έκθεση με τις τροπολογίες ε, είναι διαθέσιμη για τους διερμηνείς Επίσης, έχουμε ορισμένα αντίγραφα για τις ε, πιο συχνά χρησιμοποιούμενες γλώσσες, περίπου 120 αντίτυπα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου 6.500 σελίδες, 3,5 μέτρα χαρτιού. Εγώ προσωπικά εξοικονόμησα χαρτί γιατί είμαι ένα από τα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το iPad και την ε, ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής μας. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι και εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό εάν γραφτείτε στο σύστημα e-committee της Επιτροπής μας. Ίσως την επόμενη φορά. Οι φάκελοι αυτοί θα εκτυπωθούν μία φορά και δεν θα είναι διαθέσιμοι ξανά στην επόμενη συνεδρίαση. Τώρα να σας υπενθυμίσω ότι οι δύο επιτροπέ ε, προετοίμασαν μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία κοινά σύμφωνα με την ε, διαδικασία του κανόνα 51 του εσωτερικού κανονισμού, έτσι όπως έχει εγκριθεί από την διάσκεψη των Προέδρων στις 26 Ιουνίου του 2013. Συνεπώ οι δύο συνεισηγητέ των Επιτροπών ΕΝΒΙ και ΙΤΡΑ έχουν προετοιμάσει κατόπιν κοινή συμφωνία σε ένα κοινό σχέδιο έκθεση. Όπω σα είπα, 920 τροπολογίε υποβλήθηκαν και οι συνεισηγητέ και οι σκιώδε εισηγητές συμφώνησαν να καταθέσουν συμβιβαστικέ τροπολογίε μέχρι τι 12 Δεκεμβρίου και, πολύ σημαντικό, να θεωρηθούν συμβιβασμοί εάν υπογραφούν από τουλάχιστον τρει ε, σκιώδεις ή συνεισηγητέ. Διαφορετικά θα θεωρηθούν ως ενοποιημένες τροπολογίες. Να σας ε, υπενθυμίσω ότι στις συμβαστικές τροπολογίες δεν ε, γίνεται να τις ψηφίσουμε κατά τμήματα. Η έκθεση θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στις κοινέ συνεδριάσεις των δύο επιτροπών. Υπάρχει και ξεχωριστό σχέδιο ημερήσια διάταξη για τις κοινέ αυτές συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις αυτές ε, έχουν πάντα δύο προέδρους. Η κυρία Σαρτόρη θα έρθει σύντομα. Το αεροπλάνο της είχε μια μικρή καθυστέρηση. Τώρα, για να διευκολύνουμε την διαδικασία, οι δύο επιτροπές συμφώνησαν ότι ο πρόεδρος ότι οι δύο πρόεδροι θα συμπροεδρεύσουν. Αυτή η, επιτροπή, η συνεδρίαση θα έχει την Επιτροπή Ένβη ως πρόεδρο. Ωστόσο, και ο πρόεδρος της άλλης επιτροπής θα έχει το δικαίωμα παρεμβάσεων. Τώρα, κανονικά θα έδινα το λόγο στην κυρία Σαρτόρη, αλλά μια και θα έρθει αργότερα, δεν θα το κάνω. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 3, έγκριση των παρακτικών, συμπεριλαμβάνοντα τα έγγραφα της συνεδρίασης και αν δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρούμε την ημερήσια διάταξη, τα πρακτικά εγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ. Και με αυτό περνάμε στο σημείο 4, το πλαίσιο για το 2030 για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική. Θα αρχίσω δίνοντας ε, το λόγο στους συνεισηγητές. Η Σοφή Οκουνή, να σας ενημερώσω ότι θα αντικαταστήσει σήμερα την Αντελβό. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω δίνοντας το λόγο στον άλλο συνεισηγητή, τον κύριο Σιμάντσκι και οι δύο θα έχετε από 10 λεπτά έκαστος. Ευχαριστώ πολύ. E, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σε σχέση και με το ότι από πλευράς τώρα αυτών των τροπολογιών, από πλευράς γραμματείας που δεν ε, διατίθενται σε όλους, ε, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και εγώ θα προσπαθήσω να εξοικονομήσω ε, δεν πρόκειται τώρα προσωπικά να τοποθετηθώ σε κάθε μία από αυτές τις τόσες πολλές τροπολογίες. Θα ήθελα να πω αυτά που έχουμε μπροστά μας και είναι τα πιο φλέγοντα θέματα, σε αυτά θα ήθελα να επικεντρωθώ. Οι συμβιβασμοί είναι οι πιο σημαντικές υποθέσεις σε όλους τους τομείς. Παρότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό τροπολογιών, είναι δυνατόν να εκπονήσουμε συμβιβαστικές τροπολογίες, διότι πολλοί ευρωβουλευτές τις δικές τους ε, προτάσεις, τις δικές τους ε, τροπολογίες τις κατέθεσαν, αλλά πολλά πράγματα βαίνουν προς την μία κοινή κατεύθυνση. Γι' αυτό μπορούμε συχνά αυτές ε, τις τροπολογίες που βαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση να τις παγιώσουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Αυτό διευκολύνει τα πράγματα και έτσι μπορούμε και να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έγγραφο θα είναι εύληπτο και σαφές ε, και θα μπορεί κανείς να το κατανοήσει εύκολα και θα έχει μια σαφή γραμμή οι συμβιβασμοί προς αυτή την κατεύθυνση ε, θα εκπονηθούν. Νομίζω δύο σημαντικά πράγματα πρέπει να αναφερθούν και να ληφθούν υπόψη. Καταρχήν πρώτα θα ήθελα να πω ότι όλους τους σκιώδεις εισηγητές θα ήθελα να τους προειδοποιήσω κρουοκόδωνα κινδύνου, να μην πιστέψουν οι σκιώδεις εισηγητές ότι 50% συν 1, δηλαδή 51% σε κάποιο σημείο της έκθεσης μπορεί να ε, ρυθμιστεί έτσι. Φυσικά σε μια νομοθετική έκθεση <clears throat> με μια πολύ μικρή πλειοψηφία δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε έτσι. Και το ψήφισμα πρέπει να είναι ένα ψήφισμα του συνόλου του Ευρωκοινοβουλίου. Αν όμως δούμε την δυναμική των πραγμάτων πώς έχει εξελιχθεί σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την φωνή που πρέπει να αρθρώνει το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο για μια ευρύτερη συζήτηση έναντι για παράδειγμα του Συμβουλίου θα έπρεπε να εργαστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί πλειοψηφικά, με σημαντικό τρόπο πλειοψηφικά να εγκρίνει κάποια πράγματα. Δεν θα ήταν φιλόδοξο αν επιτρέπαμε απλά και μόνο κάποια πράγματα να περάσουν με μικρές πλειοψηφίες, με οποιαδήποτε μικρή πλειοψηφία κάποια πράγματα να πούμε. Δεν θα ήταν αυτό το πιο εύθετο. Αυτή η έκθεση πρέπει να ε, είναι, ας το πω έτσι, αποτελεσματική και θα το υπενθυμίζω διαρκώς αυτό ότι πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα μείζον πρόβλημα έχουμε ε, ενώπιον μας. Υπάρχουν φυσικά προσπάθειες, εγχείρημα που ακολουθείται να επιτευχθεί μια μικρή πλειοψηφία και να, έτσι να εγκριθεί. Αυτό θα ήταν όμως επιζήμιο για το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν κάποιοι ευρωβουλευτές από διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες που προσπαθούν από πλευράς τους, ας το πω έτσι, ε, λες και υπάρχει ε, δυνατότητα καταλήγουμε σε ε, κάποια διέξοδα διπολικού χαρακτήρα ή το ένα ή το άλλο αλλά πρέπει να δούμε θα έχουμε ένα υποχρεωτικό στόχο δύο υποχρεωτικού στόχους Νομίζω από αυτό το αδιέξοδο μπορούμε να διεξέλθουμε, να αποφύγουμε το αδιέξοδο αν είμαστε δημιουργικοί. Εφάνταστη δημιουργική προσπάθεια είναι αυτό που χρειάζεται για αυτή την έκθεση. Αν διαπιστωθεί ότι το Ευρωκοινοβούλιο για τον έναν ή άλλο λόγο θεωρεί ότι το μόνο το οποίο εδώ ως μήνυμα θα έπρεπε να σηματοδοτήσουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μόνο θα ήταν ουσιαστικά η επανάληψη αυτών που έχουν αναφερθεί κατά το παρελθόν και μάλιστα επανειλημμένα, ε τότε θα έλεγα ότι δεν θα ήταν καλό κάτι τέτοιο θα έπρεπε τη δική μας πείρα σε σχέση με τα κλιματικά θέματα να την εκμεταλλευτούμε. Δεν στρέφομαι σε κάποιο συγκεκριμένο συνάδελφο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε με κριτικό πνεύμα να φωτίσουμε τα όσα συνέβησαν και με κριτικό πνεύμα πάντα να δούμε τι πρέπει να γίνει. Έχουμε κάποια πείρα που έχουμε συλλέξει και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ένας βαθμός υψηλής ελαστικότητας, ευελιξίας Ιδιαίτερα μετά την κρίση υπάρχουν τελείως διαφορετικά αιτήματα και απαιτήσει, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χρειάζονται τρεις ε, σημαντικοί στρατηγικοί στόχοι να συνδυαστούν μεταξύ τους που από αυτό το νομοθετικό πακέτο απορρέουν. Α, καταρχήν η αηφορία στην ανάπτυξη, η ε, τροφοδότηση των ενεργειακών αναγκών μας και η ενεργειακή ανεξαρτησία. Αυτές οι τρεις κατευθύνσεις πρέπει να είναι δεδομένες και κύριες στην έκθεσή μας. Δεν είναι δυνατόν ε, να, κατέβουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο και έτσι στην νομοθετική μας δράση να έχουμε ένα πακέτο μέτρων Μία δέσμη μέτρων που δεν θα είναι ισορροπημένη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που είναι νέες και απόλυτα καινούριε. Αυτές οι προκλήσεις πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν τόσο σαφείς. Η τιμές της ενέργειας, των ενεργειακών προϊόντων για παράδειγμα και των πιο σημαντικών εταίρων μας εξάλλου. Όλοι οι πιο σημαντικοί εμπορικοί μας εταίροι εκτός από την Ιαπωνία έχουν ένα προτέρημα στον ανταγωνισμό και έχουν πολύ χαμηλές ενεργειακές τιμές, ιδιαίτερα όσον αφορά το φυσικό αέριο. Με την, τις Ηνωμένε Πολιτείε θέλουμε να υπογράψουμε την συμφωνία επενδύσεων και ε, νέων ε, δράσεων ε, ώστε να δούμε πώς θα πρικοδοτηθεί η ενεργειακή πολιτική μέσα σε αυτό το πακέτο. Θα ήταν πολύ χαμηλές οι προσδοκίες μας αν περιορίζαμε το ευρώ στο φάσμα αυτό θα πρέπει από τις διαφορετικές προσδοκίες να τις συνδυάσουμε και να τις συνδέσουμε μεταξύ τους και να είμαστε τόσο ελαστικοί και ευέλικτοι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε με αυτόν τον τρόπο στις προσδοκίες. Όπως και ο κύριος Γκεμπράντι πριν από κάποιες εβδομάδες είχε αναφέρει, αυτό που σήμερα εγώ προσπάθησα κατά τη διάρκεια της ε, μετάβασής μου προς το Ευρωκοινοβούλιο σήμερα μελέτησα την εφημερίδα Financial ε, Times και είδαμε τα θέματα, είδα τα θέματα του πακέτου 2030 και θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με ε, ακριβούς ενεργειακούς στόχους για το 2020 διακυβεύουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί να επαναλάβουν ε, τα ίδια λάθη με, ένα νέο, ε, με νέους στόχους στο εγχείρημά τους. Τα επανειλημμένα λάθη της προηγούμενης δεκαετίας θα μπορούσαν έτσι να επιβιώσουν σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Και αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη ανοησία όλων. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι σε αυτό αναφέρεται στην Financial Times. Και βλέπουμε ότι δεν συμφωνώ πάντα βέβαια με τα όσα λέει η Financial Times, αλλά σε αυτή την περίπτωση συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Ένας αριθμός τροπολογιών αντανακλά αυτή την δημιουργική τοποθέτηση, δημιουργικό προβληματισμό. Βλέπουμε ότι αυτή η εφάνταστη δημιουργική ε, δράση στη σκέψη μας ε, μπορεί να βρει ε, απήχηση και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Άρχισε να ανεβαίνει ο ήχος όταν κάνατε τις τελικές σας παρατηρήσεις. Ωραίο κόλπο αυτό. Αντικαθιστώντας την άλλη εισηγήτρια, έχει το λόγο η κυρία Οκονή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε, η Αντολβό, η συνεισηγήτρια, για ιατρικούς λόγους δεν είναι σε θέση να είναι παρούσα και μου ζήτησε να την αντικαταστήσω. Την ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη της και της εύχομαι εκ μέρους όλων καλή ανάρρωση. Όλοι είστε γνώστες των 920 τροπολογιών που κατετέθησαν και θα ήθελα εξ ονόματος της Ντολβό να σας ευχαριστήσω όλους γιατί προσπαθήσατε να εμπλουτίσετε την έκθεση. Βλέποντας τόσες πολλές τροπολογίες είδα ότι τελικά συμμεριζόμαστε τους στόχους, τους γενικούς στόχους. Είμαστε υπέρ μιας ανταγωνιστικής, ενεργειακά ανεξάρτητης Ευρώπης, και με μια οικονομία που θα αναπτυχθεί με αηφορία σεβόμενη τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Βέβαια διαφέρουν τα μέσα για να πετύχουμε αυτούς τους γενικούς στόχους. Από την αρχή των εργασιών φαίνεται ότι υπάρχουν δύο οράματα παράλληλα στο εσωτερικό της Επιτροπής μας καταρχάς ε, ε, δεσμευτικές μειώσεις στις εκπομπές που αφήνει ε, μια κάποια άνεση στα κράτη-μέλη για τους τρόπους και για το πότε. Και από την άλλη υπάρχει μια αντίληψη που προτείνει ορισμένες τεχνολογίες αναγνωρισμένες ως χρήσιμες και που αξιολογεί τις πολιτικές που έχουν ήδη ξεκινήσει όπως οι επενδύσεις στα ανανεώσιμες πηγές και στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πρώτη διαφορά. Χαίρομαι γιατί διαπιστώνω πάντως μέσω των τροπολογιών σας την συγκεκριμενοποίηση για την στήριξη την οποία διείδαμε και στην προηγούμενη συζήτηση γύρω από το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπει κανείς ότι αναγνωρίζονται τα μεγάλα πλεονεκτήματα που μια σωστή πολιτική μπορεί να προσφέρει στον τομέα της μείωσης του κόστους χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος, στα πλαίσια της μείωσης της γενικότερης ενεργειακής δαπάνης και στα πλαίσια της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης μονίμων τοπικά, μη μετακινήσιμων. Στόχος 40% βελτίωση αποδοτικότητας μέσα σε 10 έτη. Η καλύτερη τροχιά θα μας επιτρέψει να μειώσουμε κατά 50% ε, τις εκπομπές ε, καυσαερίων θερμοκηπίου και να αυξήσουμε κατά 40% το ποσοστό των ανανεώσιμων στη ε, μίξη, στο μείγμα ενεργειών που χρησιμοποιούμε. Όμως η πιθανή συγγραφή στη συγκεκριμένη περίπτωση συμβιβαστικών τροπολογιών δεν μπορεί παρά να λάβει υπόψη τις αντιθέσεις αυτές. Πόσοι στόχοι σαν παράδειγμα θα πρέπει να υπάρχουν. Θα πρέπει άραγε ε, να υπάρχει ένας δεσμευτικός χαρακτήρας και σε ποιο επίπεδο. Ελήφθη η απόφαση με τους κοιόδης εισηγητές ότι κάθε πρόταση η οποία θα συνυπογραφεί τουλάχιστον από τρεις σκιώδεις εισηγητές ή συνεισηγητές θα θεωρηθεί συμβιβαστική τροπολογία. Μπορείτε να φανταστείτε ότι με δύο συνεισηγητές και δώδεκα σκιώδεις εισηγητές οι πιθανότητες εδώ συμβιβαστικών είναι πολλαπλές. Πέραν των ακαθοδών αν θέλετε θεμάτων υπάρχουν και πολλές συγκλήσεις. Αναφέρομαι στο κεφάλαιο για την συνεκτικότητα των μέσων, την ενεργειακή ασφάλεια, η διασφάλιση και την ανταγωνιστικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των συνεισηγητών και των σκιωδών και των ομάδων τους που έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια ισόρροπη και ευκρινή έκθεση και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο σε αυτό το πλαίσιο να μου επιτρέψετε να μπω σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει αρκετή συνένεση για να πούμε ότι απαιτείται περισσότερη συνεκτικότητα στις εθνικές πολιτικές στήριξης ανεξαρτήτως της κάθε φορά ε, χρησιμοποιούμενης μορφής ενέργειας. Για το 2003 πρέπει να αποτύχουμε τα λάθη του προηγουμένου χρονικού πλαισίου, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη όλες τις μορφές αλληλοεπιδράσεων και αλληλοεπιρροών που κάθε μέτρο στο εσωτερικό του πλαισίου θα έχει εις βάρος των υπολείπων μέτρων, ιδιαίτερα στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και ένα μακροπρόθεσμο όρεμα που να συνοδεύεται από ένα σταθερό και ξεκάθαρο διακανονιστικό πλαίσιο που να προσφέρει ασφάλεια στις επενδύσεις και του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Νομική ασφάλεια, διακανονιστική ασφάλεια πρέπει να είναι βασικός μας στόχος. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε επίσης τις διασυνδέσεις δικτύων ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να βελτιστοποιήσουμε το ενεργειακό μίξ και να χρησιμοποιήσουμε κυρίως τις ενέργειες, την ενέργεια συγγνώμη, που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι κανόνες στον τομέα της αποδοτικότητας μπορούμε μέτρα να πάρουμε όπως τις μεταφορές ή τις κατασκευές μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητη ανάμεσα στα κράτη-μέλη όταν λαμβάνονται στρατηγικού τύπου εθνικές αποφάσεις, οι οποίες όμως έχουν συνέπειες στις γειτονικές περιοχές και χώρες. Είναι απαραίτητο για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας και την ανταγωνιστικότητα των εταιριών μας να προλαμβάνουμε επίσης και τους κινδύνους διαφυγής διοξιδίου. Πρέπει να βελτιώσουμε και να καταστήσουμε αποδοτικότερη την πρόσβαση στην χρηματοδότηση που θα υποστηρίξει τις τεχνολογίες στις αηφόρες τεχνολογίες ευρωπαϊκής κλίμακας Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας, έχουμε πολύ υλικό έτσι ώστε να εκφραστούμε με συγκεκριμένο τρόπο, με ευκρινή τρόπο και να επηρεάσουμε συγκεκριμένα το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την θέση που έχει στην διεθνή σκηνή. Πριν κλείσω θα ήθελα να κάνω έκκληση στον καθένα σας να χρησιμοποιήσετε το πνεύμα το συμβιβαστικό που μπορεί να σας διέπει για να βρούμε λύσεις το απτό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Δεν πρέπει να αγνοούμε την πραγματικότητα, πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον τομέα των στρατηγικών προσανατολισμών. Θα ακούσω με ενδιαφέρον τις απόψεις σας και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με αυτές τις τροπολογίες τις οποίες θα μεταφέρω στην κυρία Ντολβό. Ευχαριστώ πολύ κυρία ακούνη να μεταφέρετε και στην ε, κυρία Ντελβό τις ευχές μας για καλή ανάρρωση και γρήγορη ανάρρωση. Τώρα, περνάμε στους ασκαιώτες εισηγητές. Είναι μακρύς ο κατάλογος, δεν είναι όλοι παρόντες. Προτείνω λοιπόν να ακολουθήσουμε την, ε, τον, τη σειρά με την οποία έχω τους ασκαιώδες εισηγητές στον καταλογό μου. Προτείνω πέντε λεπτά χρονομιλίας για τον κάθε ασκαιώδη εισηγητή και αρχίζουμε με τον κύριο Χέρμπερτ Ρόιλ εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Αν και δεν ζήτησα το λόγο. Καταρχάς, να πω ότι φυσικά οι τροπολογίες είναι πάρα πολλέ και η δουλειά μας είναι να φροντίσουμε να μην παραλείψουμε πράγματα. Να προσέξουμε επίσης ε, να ε, συγκεντρώσουμε τις ε, παρόμοιες τροπολογίες και να μην παραβλέψουμε τις ε, διαφορές. Είναι φυσιολογικός τρόπος αυτός λειτουργία σε μια δημοκρατία. Δεν μπορούμε και δεν χρειάζεται να εξετάσουμε παρόμοια πράγματα. Είναι όμω πολύ ε, σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτά τα πράγματα που εμεί θεωρούμε πολύ σημαντικά και που είναι πολιτικά σημαντικά. Πάντα γίνεται λόγος ε, για το ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο φιλόδοξοι. όμω όσο πιο πολύ το ακούω τόσο πιο ε, λίγα πράγματα έχω να πω γιατί ακούμε συνέχεια για φιλοδοξία. Αλλά Όσον αφορά την ε, προστασία του περιβάλλοντος ε, στην Ευρώπη, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει και εκπληκτική πρόοδο. Ε, πραγματικά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Θέλουμε μεν να επιτύχουμε τους στόχους, όμως διαθέτουμε πολύ λίγα κονδύλια και αναλογικά αυτό δεν ευσταθεί. Πρέπει καταρχάς να δούμε εάν ο τρόπο, η μέθοδο, τα μέσα που διαθέτουμε είναι τα σωστά για να το αντιμετωπίσουμε, εάν τα μέσα αυτά είναι αποτελεσματικά ή αν πρέπει να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό. Περισσότεροι στόχοι, ψηλότεροι στόχοι, όλο ένα και περισσότερη τελειομανία. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε διαφορετικά το θέμα. Ελπίζω να πω να μην συγκρουστούμε να μην συγκρουστούν οι απόψεις μας. Ελπίζω να έχουμε πραγματικά το χρόνο να δούμε τα πράγματα, να τα συζητήσουμε και να δούμε εάν είναι η μέθοδος που ακολουθούμε η καλύτερη, αν πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική προσέγγιση. Διότι στην Ευρώπη χρειαζόμαστε νέες θέσεις εργασίας, χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Αυτή είναι οι τομή στους οποίους δυσκολευόμαστε. Άλλες χώρες περισσότερο, άλλες χώρες λιγότερο. Έχουμε πραγματικά ένα υπαρκτό πρόβλημα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και κάνουμε πράγματα γι' αυτό, όχι όμως τόσα όσα θα θέλαμε και όσα θα έπρεπε. Πρέπει να προσέξουμε το κόστος της ενέργειας, το οποίο ε, είναι απαγορευτικό για πάρα πολλούς και οδηγεί σε οριακές καταστάσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα αυτό με περισσότερες προδιαγραφές ή με πιο έξυπνη αντιμετώπιση, με διαφορετική αντιμετώπιση. Γι' αυτό πιστεύω και μπορώ να μιλήσω και εκ μέρους του συναδέλφου Ρόμαν Γιόρταν, ο οποίος λείπει και μου ζήτησε να μιλήσω εκ μέρους του. Πιστεύω λοιπόν ότι ο σωστός ο τρόπος είναι να επικεντρωθούμε στον πιο σημαντικό στόχο. Να δούμε τα μέσα. Να δούμε τα μέσα και πώς αυτά μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Να δούμε αν λειτουργεί πραγματικά το σύστημα εμπορίας εκπομπών και αν λειτουργεί αποτελεσματικά. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών ένα μέσο αποτελεσματικό και να επεξεργαστούμε παράλληλα και τους άλλους ε, στόχους. Τους τελευταίους μήνες έχουμε αντλήσει διδάγματα. Έχουμε δει ότι ε, όταν υπάρχουν ε, αντίθετοι παράλληλοι στόχοι δεν βοηθούν στο να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Και αυτό έγινε και με το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Και πραγματικά αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας θα δούμε και το πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα δούμε πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χαμηλότερο, με προσιτό κόστος. Πρέπει πραγματικά τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τους εγωισμούς τους και να συγκεντρωθούν σε μια κοινή λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό. Πώ λοιπόν θα προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια ε, στο μέλλον, πώς θα τις αναπτύξουμε. Διαφορετικά δεν θα πάμε μπροστά και εύχομαι να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση, να ακολουθήσουμε αυτόν τον κοινό δρόμο, να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο κόστος, χαμηλότερο ε, βάρος ε, προς τους ε, πολίτες, με όσο το δυνατόν λιγότερα μέσα, λίγα και αποτελεσματικά, λίγα και καλά. Αυτά είχα να πω στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρόιλ. Περνάμε στην κυρία Ούλσκοκ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως αυτό που πρότεινε ο κύριος Ρόιλ είναι καλό. Χρειάζεται να τονιστεί η σημασία των συμβιβασμών. Γιατί? Διότι Εάν δεν είμαστε σε θέση να συμβιβαστούμε, αν δεν πάρουμε τους συμβιβασμού στα σοβαρά, δεν θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε το έργο μας. Εμείς ως θεσμικό όργανο, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστούμε και τις συνέπειες της άρνησής μας αυτής. Σίγουρα, για μένα τουλάχιστον, και για την ε, κοινοβουλευτική μου ομάδα πρέπει να ε, αφαιρέσουμε τη λέξη φιλοδοξία, φιλόδοξος από τα διάφορα σημεία της ε, έκθεσης. Είναι κάπως προκλητική αυτή η διατύπωση, αν το δούμε από διαφορετική σκοπιά και θα σας ε, πω και γιατί. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Στην τροπολογία 231 του ΕΛΚ αναφέρεται ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές δεν είναι λιγότερο σημαντικές από άλλες ε, πολιτικές, σε άλλους τομείς. Αυτή η δήλωση τουλάχιστον για ορισμένου από εμάς, ε, είναι προκλητική. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αφαιρεθεί, πρέπει να αφαιρεθεί αυτός ο προκλητικός χαρακτήρας της ε, διατυπώσεις φιλόδοξου. Μετά, τροπολογία 290 του ΕΛΚ. Και αυτό είναι προκλητικό για πολλούς από εμάς διότι αναφέρεται ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να θέσουμε περιβαλλοντικούς στόχους αφότου καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και δηλαδή δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτό που κάνουμε είναι, είναι θεραπεία, είναι αντιμετώπιση. Ότι δηλαδή θα δράσουμε του λήξει η συμφωνία για να δημιουργήσουμε μια νέα συμφωνία. Και αυτό είναι προκλητική δήλωση. Εντάξει, παραδέχομαι ότι και από τη δική μας πλευρά θα υπάρχουν στοιχεία που οι άλλοι θα θεωρήσουν προκλητικά, αλλά πρέπει να συμβιβαστούμε έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια συνετή και λογική αποδεκτή λύση για όλους. Πρέπει να συζητήσουμε για αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε και να μην εισέλθουμε σε μάχη για τις επιμέρους τροπολογίες. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία είναι ξεκάθαρα, τουλάχιστον ε, για εμάς τους σοσιαλδημοκράτες. Και είναι θέσεις ε, τις οποίες είχαμε ευθύς εξ αρχής. Θέλουμε τρεις στόχους. Μείωση των εκπομπών, δημιουργία περισσότερων ανανεώσιμων και αποτελεσματικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και θέλουμε να είναι δεσμευτική αυτή η στόχη. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στόχος ενεργειακής απόδοσης, δεν είναι όμως δεσμευτικός και γι' αυτό δεν έχουμε καταφέρει τόσα όσα θέλαμε, ιδιαίτερα ε, σε σχέση με τους ε, άλλους ε, δύο δεσμευτικούς στόχους. Αυτό που επίσης επιθυμούμε είναι ξεκάθαρα νούμερα όσον αφορά τα, τους στόχους της ε, κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής. Ξεκάθαρα νούμερα. Και όσον αφορά τα νούμερα αυτά, τους στόχους αυτούς, να πω ότι δεν τους θεωρούμε αρκετά υψηλούς. Επίσης, τουλάχιστον η δική μου ομάδα είναι έτοιμη να συνεργαστεί όσον αφορά τις τιμές. Όμως αυτό να το δούμε ως ε, αποτέλεσμα, ενδεχομένως ως κανονισμό σχετικά με την εμπορία εκπομπών. Και επίσης δεν είναι πιστεύω σωστό να ψάχνουμε ποιος φταίει Ποιος έφταιγε που δεν λειτουργήσε το σύστημα. Όχι, α αφήσουμε κατά μέρου όλα αυτά τα παιχνίδια. Ας μην προσπαθούμε να βρούμε το μαύρο πρόβατο. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα βγει κάποιος από πάνω. Δεν πρέπει να δαχτυλοδείχνουμε. όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ήταν εντάξει και αυτό που χρειάζεται είναι βελτίωση. Και την ευκαιρία την έχουμε, την έχουμε εδώ, την έχουμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η παιδιάστικη συζήτηση και διαφωνία που έχουμε δεν έχει νόημα. Για εμάς λοιπόν σημασία έχουν τρεις στόχοι, δεσμευτικοί, με σαφή νούμερα, σαφείς τιμές και μετά ας συζητήσουμε για τον κανονισμό του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τα πράγματα περίπλοκα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ροτσκόκ. Και ιδιαίτερα ορίζοντας την κυρία Σαρτόρη, δίνω το λόγο εξ ονόματος ε, της ε, Άλντε, παρακαλώ για να παρέμβετε. Σας ευχαριστώ. Σημείωσα ότι πολλές από τις τροπολογίες που έχουμε εδώ αφορούν την ανταγωνιστικότητα και ελπίζω ότι είναι σημεία επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε ως κοινά σημεία. Έχουμε και κάτι επί από το οποίο δεν μπορούμε να διαφύγουμε επειδή φυσικά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προετοιμάζει τις προτάσεις της και πρέπει να καταθέσουμε και εμείς τις δικές μας απόψεις Θέλω να δραθώ τις ευκαιρίες και να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες και όλους που εργάστηκαν σκληρά σε τεχνικό επίπεδο για να εξευρεθούν συμβιβασμοί για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Με χαρά σκέφτηκα πόσες τροπολογίες τονίζουν πόσο απαραίτητη είναι η αποδοτικότητα στην εκμετάλλευση της ενέργειας για την αποτελεσματικότητα γενικά και όσον αφορά και τα θέματα ασφάλειας από την EIA που τονίζεται ότι πρέπει να εξετάζεται η αποδοτικότητα της ενέργειας ε, πρώτα και κύρια Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα χρονολογικό ζήτημα όσον αφορά την οδηγία για την αποδοτικότητα και την αναθεώρηση η οποία δεν έχει γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Θα πρέπει όμως αυτή την έκθεση να προβληματιστούμε και να δούμε πόσο κέρια σημασία και σπουδαιότητα έχει το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας ελπίζοντας ότι πολλοί συνάδελφοι από διαφορετικές ομάδες θα καταθέσουν και θα τοποθετηθούν με ένα αποτελεσματικό, ε, μια αποτελεσματική αναλογία σε σχέση με τις τιμές ώστε να έχουμε μείωση κατά 40% ως ε, μέχρι το 2030 και εδώ πολλά μπορούν να γίνουν και όσο αφορά και τις μεταφορές ε, αισθάνομαι ότι έχουμε το δυναμικό να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή γλώσσα και ορολογία για ένα στεναρό, μια στεναρή επικέντρωση σε θέματα φιλόδοξων στόχων όσον αφορά την αποδοτικότητα της ενέργειας. Θα πρέπει πραγματικά να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται λόγος για τα αέρια του θερμοκηπίου και πολλές φορές μπορεί να γίνει πολύ πιο δαπανηρή η μείωση του άνθρακα. Θα πρέπει να κάνουμε εκείνο το οποίο είναι το πιο αποτελεσματικό από πλευράς μας, γιατί διαφορετικά θα καταλήγουμε όλο και περισσότερο στην εμπορία ρήπων και έτσι θα έχουμε μικρότερες επιδόσεις. Βέβαια πάντα με την αρχή ότι ο ρηπαίνων πληρώνει. Τώρα, για μεγάλη αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας που πρέπει να μπορεί να μεταφράζεται σε σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ακόμα και ως 50% για τα ανανεώσιμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την αποσύνδεση του θέματος ε, του ενεργειακού κόστους ε, και την υποστήριξη των ανανεώσιμων για την ανάγκη να προαθούν τα ανανεώσιμα για τις ενεργειακές τιμές πολλές πληροφορίες βρίσκονται σε κυκλοφορία. Όλες οι αναλύσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη δείχνουν ότι οι τιμές των ορυκτών καυσίμων και μάλιστα σε σχέση με, τα, με τις ανανεώσιμες πηγές ε, ε, ενέργειας πληρώνουμε πολύ περισσότερο για τα ορυκτά καύσιμα και θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι Πρέπει να ε, ε, ξαναδούμε τα θέματα των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να συναγάγουμε τα σωστότερα συμπεράσματα. Αλλά πρέπει να μην συγχέουμε τα θέματα αυτά με τη σπουδαιότητα των ανανεώσιμων. Και αυτό επειδή πρέπει να έχουμε ένα στόχο για τα ανανεώσιμα πέρα από τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Πρέπει να βρούμε και να θέσουμε ε, τέτοιου είδους κίνητρα από πλευράς ε, ETF, ώστε αν θέλουμε να προαγάγουμε τις επενδύσεις για τα ανανεώσιμα μέσω του συστήματος εμπορίας ρήπων, να δούμε πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Το δεύτερο, να μην υπάρχει αβεβαιότητα σε σχέση με τα ανανεώσιμα που μπορεί να αυξήσει το κόστος. Μας λένε οι επενδυτές, αν γνωρίζουν, αν μπορούν να γνωρίζουν ότι θα προαχθούν σε συγκεκριμένο ποσοστό τα ανανεώσιμα, αυτό μειώνει το κόστος της επένδυσης, το καθιστά λιγότερο δαπανηρό. Πρέπει να γνωρίζουν και να ξέρουμε τι κάνουμε για να μπορέσουμε να προαγάγουμε τα ανανεώσιμα μέχρι το 2050 με ε, τον πιο φιλόδοξο στόχο να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τα αέρια θερμοκηπίου. Να μην υπάρχει υψηλότερο κόστος για τα ανανεώσιμα, πράγμα το οποίο θα τα επιβαρύνει. Συνοψίζοντας θα ήθελα να πω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε αξιολογώντας τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να πετύχουμε το κόστος ενέργειας που θα είναι πιο αποδοτικό για τα ανανεώσιμα και να θέσουμε στόχους με βάση αυτή τη διεργασία και ελπίζω ότι σε σχέση με τις τροπολογίες θα μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία επ' αυτών πώς θα κινηθούμε. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να δούμε την ανταγωνιστικότητα και την δυνατότητα της προώθησης της ανάπτυξης ανεξάρτητα και να μην χωλένουμε και βρεθούμε ουραγοί πίσω από άλλες ε, χώρες ε, και σε σχέση με την προαγωγή από αυτούς τα, των ανανεώσιμων να βρεθούμε εμείς ε, ως ουραγοί και να μην μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Τρίτο και ολοκληρώνω, πρέπει να θυμόμαστε πάντα πώς αλλάζουν τα πράγματα και σε σχέση με το Συμβούλιο έχουμε και σε σχέση με τη Γερμανία, Ομοσπονδιακή Γερμανία, την προοπτική μιας νέας κυβέρνησης και πρέπει να δούμε αυτή την προσέγγιση και για την μετάθεση του κέντρου βάρους του στο Συμβούλιο πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλοι ε, από πλευράς ε, δεν έχω πολλά να προσθέσω ως ε, σκιώδης εισηγητής και δεν θα ήθελα να αποδυναμώσω τον φιλελεύθερο, ε, την φιλελεύθερη αισιόδοξη αυτή νότα την οποία παρουσιάσατε. Έχουμε και έναν κατάλογο εδώ ενώπιον μας. Ο επόμενος είναι ο κύριος Σιμάνσκι για τον γύρο μετά τους σκιώδης εισηγητές. Έχουμε μόνο έναν ευρωβουλευτή που ζητεί να παρέμβει τον κύριο Ιβο Πίλετ, την κυρία Χέρτσοκ. Αν υπάρχουν άλλοι ευρωβουλευτές που θέλουν να παρέμβουν, παρακαλώ να μου το γνωστοποιήσετε. Ο κύριο Σιμάνσκι έχει τώρα τον λόγο, παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, Επ' αυτού θα ήθελα να πω το εξή. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί ένα συμβιβασμό. Δύσκολο το έργο αυτό. Γιατί? Διότι όταν μιλάμε για μια θεραπεία πρέπει πρώτα να υπάρξει διάγνωση της ασθένεια. Πώ έχει η κατάσταση για παράδειγμα και νομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Σήμερα είναι επίκαιρο, εξακολουθεί να έχει επίκαιρη σπουδαιότητα σε σχέση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από το 2008 διότι αυτά τα οποία αναφέρθηκαν το 2008 είναι επίκαιρα σήμερα. Έχουμε εδώ το στόχο για παράδειγμα για το 2020 και τα κράτη-μέλη με διαφορετικό τρόπο θέλουν να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους. Υπάρχουν προβλήματα από κράτη που έχουν περάσει μέσα από μια διαδικασία μετάβασης και προσαρμογής Γίνεται λόγος για φιλόδοξους στόχους όταν αναφέρεται η μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Φιλόδοξο κάτι μπορεί να είναι όταν όλοι συνενώνουν τις προσπάθειές τους και ακολουθούν αυτή την πορεία. Και οι μεγαλύτεροι ρήπαντες, η ΙΠΑ, η Κίνα, τότε έχει νόημα να γίνεται λόγος για κάτι τέτοιο. Και όταν και η μείωση του διοξιδίου του άνθρακα είναι σε ίδια εμβέλεια και μέτρο όπως και από δική μας πλευράς. Εναντι τίνος μου μπορεί να γίνει αυτό. Ο συμβιβασμός, για παράδειγμα, ως όταν προαναφέρθηκε η αποδοτικότητα της ενέργειας, ιδιαίτερα σημαντικός στόχος και χαμηλές ενεργειακές τιμές για τους τελικούς καταναλωτές, για τους χρήστες. Η κοινωνική διάσταση, για παράδειγμα. Βλέπουμε να υπάρχει μια δυνατότητα συμβιβασμού, αλλά αυτά τα οποία ακολουθούν θα πρέπει να οδηγήσουν σε περαιτέρω μειώσεις. Πρέπει όμως να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και πρέπει να προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε και φοβούμε ότι όταν τα ουσιοδέστερα πράγματα δεν τα έχουμε εγκρίνει και δεν έχουμε προχωρήσει, δεν μπορούμε να καταλήγουμε σε συμβιβασμούς. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ήδη σήμερα, για παράδειγμα, στην Ευρώπη υπάρχει μια μετάθεση επιχειρήσεων και βιομηχανιών μετατίθενται και μετεγκαθίστανται εκτός Ευρώπης οι βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ε, πλήγμα και πολύ σημαντικός κίνδυνος, διότι όταν πηγαίνουν στην Κίνα ή στις ΗΠΑ τέτοιες επιχειρήσεις τότε ακόμα περισσότερες εκπομπές ρήπων, δηλαδή διοξιδίου του άνθρακα, επιτυγχάνονται. Και είναι και ένα πλήγμα κατά της δικής μας αγοράς εργασίας. Χάνουμε θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν την οικονομική συνιστόσα και όλες οι τροπολογίες θα πρέπει υπό το φως της ανταγωνιστικότητας να εξετάζονται. Ο κύριος Σιμάσκης σωστά τα ανέφερε. Οι ενεργειακές τιμές είναι πολύ διαφορετικές ε, στα διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί βιομηχανικοί τομείς ε, απλά από τις ενεργειακές τιμές εξαρτώνται. Και ξέρουμε τι γίνεται για παράδειγμα με την Ουκρανία σήμερα και ποιες επιπτώσεις έχουν όλα αυτά και ποιες ήταν, ποια ήταν η γραμμή αφετηρίας για την Ουκρανία με την απελευθέρωση για παράδειγμα της αγοράς ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Ε, λοιπόν, αυτή η προϋπόθεση που με μεγάλη δυσκολία μπορεί να υλοποιηθεί. Ναι, δεν, έχει, δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουκρανία, όμως η ενεργειακή αγορά και οι ενεργειακές τιμές για τους τελικούς χρήστες σε πολλές χώρες ήδη σήμερα είναι τόσο υψηλές αυτές οι τιμές που είναι ε, δύσκολο μπορούν να τις ανεχθούν και να τις επομισθούν ε, οι χρήστες. Και να πούμε ότι κάτι τέτοιο είναι κιόλας και φιλόδοξο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Σιμάνσκι. Περνάμε στους επόμενους ομιλητές οι οποίοι ζήτησαν το λόγο. Τρεις επιπλέον έχουν ζητήσει το λόγο. Μπελέτ, Herzog, Πρόντι. Θα ξεκινήσω με τον Μπελέτ. Ευχαριστώ πρόεδρε και οι δύο πρόεδροι μάλλον. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε μια τροπολογία που υπέβαλα μαζί με άλλους συναδέλφους. Η πιο σημαντική από αυτές τις τροπολογίες ε, είναι η 821 η 821 έχει σχέση με την διαρροή ε, άνθρακα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει τεθεί επανειλημμένα προς συζήτηση. Η συγκεκριμένη αυτή τροπολογία δεν, είναι, δεν συνιστά καινοτομία. Πρόκειται για μια ιδέα που έχει ήδη διατυπωθεί στο παρελθόν από πολλούς εμπειρογνώμονες. Υπάρχει ακαδημαϊκή έρευνα διαθέσιμη η οποία την προωθεί. Αφορά την, τον λεγόμενο φόρο BTA. Εγώ θα το ονόμαζα αυτό σαν τέλος ε, οριακών ε, ρυθμίσεων. Ε, η προσπάθεια είναι να καταστήσουμε συμφέρουσα την μεταφορά και την επεξεργασία αυτών των προϊόντων και να αντισταθμίσουμε το κόστος των φόρων που επιβάλλεται για την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Οι εξαγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξάγουν τα προϊόντα τους σε επιχειρήσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις εξαγωγές αυτές θα μπορούσαν ίσως να την χάνουν μιας κάποιας αποζημίωσης. Ως εκ τούτου λοιπόν... Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε ότι ένας, ε, ένα τέτοιο τέλος για παράδειγμα θα πρέπει να είναι συμβατό και θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει υπό την ομολογία και νομοθεσία του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Γιατί σε περίπτωση που δεν γίνεται αυτό δεκτό, και μας λέει η νέα έρευνα ότι θα μπορούσε ένα τέτοιο τέλος ε, χωρίς διακριτική μεταχείριση να λειτουργήσει αν το τέλος ε, ε, εισπράτεται από τα προϊόντα και σε σχέση με την άμεση καταβολή από τους, για παράδειγμα, τους χρήστες και θα ήθελα για παράδειγμα με το ε, Marshall Fund στην ε, Washington να ληφθεί υπόψη αυτή η τοποθέτηση και πρέπει να ευθυγραμμίζεται και με την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την εργασία η φορολογία να μετατίθεται στην ρήπανση του περιβάλλοντος και στα περιβαλλοντικά μέτρα. Αυτό προτείνουμε σε αυτή την τροπολογία. 821. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσεκτικά να εξετάσει τις δυνατότητες σε αυτό το πεδίο με βάση τη νέα πανεπιστημιακή έρευνα και για παράδειγμα την βιωσιμότητα πιλωτικών προγραμμάτων ιδιαίτερα όσον αφορά τον ενεργειακά έντονο, την ε, ε, έντονη ε, εκμετάλλευση, εντατική εκμετάλλευση ενέργειας από πλευράς βιομηχανιών. Και να δούμε σε σχέση με τις μη ευρωπαϊκές βιομηχανίες την ανάγκη να αυξηθούν οι προσπάθειες ώστε να μειωθεί ο άνθρακας, η εκπομπή άνθρακα και διοξιδίου του άνθρακα και ταυτόχρονα να υπάρξει επένδυση σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες. Θα ήθελα να έχουμε την υποστήριξη όλων των μελών α, για αυτή την τροπολογία 821. 821 <clears throat> που αναφέρεται επίσης και στις αιτιολογικές σκέψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπέλετ. Edith Herzog, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Κοιτάζοντας τις ε, διάφορες τροπολογίες Βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει σε πολλά ενεργειακά θέματα. Ότι οι δύο πλευρές ε, έχουν πιάσει τα δύο άκρα των απόψεων. Και αυτό λοιπόν θεωρώ πως θα είναι λίγο δύσκολο να οδηγηθούμε σε έναν συμβιβασμό. Είναι όμως αναγκαίος ένας τέτοιος συμβιβασμός. Διότι συμφωνώ απόλυτα με όσους ε, είπαν ότι χρειάζεται μια κατεύθυνση βασισμένη σε αυτή την άσκηση του 2013. Εγώ απέφυγα να υποβάλω τροπολογίες, θα κοιτάξω να βρω εκείνες που με αντιπροσωπεύουν, θα ήθελα όμως να σταθώ σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι αυτά που χρειάζεται να επιτευχθούν για το 2030, όποιοι στόχοι και αν είναι αυτοί, πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με τη γνώση που έχουμε, διότι η ενέργεια είναι μια πρώτη ύλη. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες γνώσεις είναι ο τρόπος ε, δημιουργίας ενέργειας. Χρειαζόμαστε λοιπόν εμπειρογνωμοσύνη, γνώση έτσι ώστε να έχουμε τους κατάλληλους συνεργάτες που θα βοηθήσουν. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν σημείο που θα κοιτάξω να βρω στις τροπολογίες. Έπειτα, θα ήθελα να αναφέρω την ανταγωνιστικότητα. Πάρα πολλοί μιλούν για ανταγωνιστικότητα και ενέργεια. Όμως τι εννοούμε. Εννοούμε την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τομέα καθ' αυτού. Και εάν ναι, τι περιμένουμε να επιτύχουμε. Τι καταλαβαίνουμε δηλαδή με τον όρο ανταγωνιστικότητα. Ορισμένοι μπορούν να το εκλαμβάνουν αυτό σε ανάπτυξη. Όμως, αν δούμε γενικά τον τομέα της βιομηχανίας, όχι μόνο της ενέργειας, ε, το... από το 2004 που ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης αντιπροσωπεύει το 30% αντιπροσώπευε το 2004 το 30% του ΑΕΠ. Τώρα τον Νοέμβριο φέτος το 15,2%, δηλαδή το μισό. Τι λοιπόν ονομάζουμε εμείς ανταγωνιστικότητα και αν το ψάξουμε ακόμα περισσότερο θα δούμε ότι αυτό το 15,1% είναι συνδεδεμένο με την ενέργεια. Και όχι μόνο με έναν τομέα. Εμείς εδώ συζητούμε επιμέρους τομείς. Την βιομηχανία χάλιβα για παράδειγμα, μετά ε, την βιομηχανία ε, αυτοκινήτων. Τα τελευταία όμως δέκα χρόνια γεγονός είναι ότι η παραγωγή έχει μειωθεί από το 30% στο 15%. Φυσικά μπορεί να το δει κανείς αλλιώς. Μπορεί να πει ότι οι υπηρεσίες έχουν αυξηθεί και έχει μειωθεί λοιπόν η ενεργειακή παραγωγή. Όμως εγώ ρωτώ, τι θα κάνουμε τώρα που μειώνεται η ενεργειακή μας παραγωγή. Τώρα, μια που μιλάμε για χάλιβα, υπάρχουν απόβλητα χάλιβα και αυτά τα απόβλητα εξάγονται στην, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μόνο το 5% του χάλιβα επαναχρησιμοποιείται. Αυτά για μια Ευρώπη που είναι ενεργειακά ανεξάρτητη ή που χρειάζεται να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη όπως λέτε. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε σαφείς ορισμούς της ανταγωνιστικότητας. Χρειάζεται σταθεροποίηση, χρειάζεται ανάπτυξη, τι απ' όλα. Ελπίζω να έχουμε μεγάλη συμφωνία, μεγάλη πλειοψηφία. Όμως, ε, συνάδελφοι, η επιτυχία δεν έγκυται στην μεγάλη μας πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Η επιτυχία έγκυται στις επενδύσεις του βιομηχανικού τομέα. Και αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε μια αναγέννηση, μια αναζωογόνηση του κλάδου αυτού, γιατί μόνο έτσι θα δημιουργηθεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Ελπίζω λοιπόν οι συγητές και οι σκιώδες συγητές να κοιτάξουν όχι τους συμβιβασμούς, αλλά το στόχο της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χέρτσογκ. Ο Βιτόριο Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Βρισκόμαστε αν θέλετε στην πέμπτη έκδοση της έκδοσης του, ε, της, του εγγράφου συγγνώμη, του International Panel for Climate Change και είναι σαφές πλέον ότι έχουμε να κάνουμε με παραγωγή και με εκπομπές ε, ε, αερίων που δημιουργεί ε, άμεσες συνέπειες μεταξύ των οποίων την υπερθέρμανση του κλίματος. Πρέπει λοιπόν σήμερα να αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε μία κάποια πρακτική πειθαρχημένα που θα μειώσει στη μείωση των εκπομπών αυτών. Βέβαια, εγώ πλέον αρχίζω να έχω αμφιβολίες για το εάν το πρωτόκολλο του Κιώτο μπορεί να βοηθήσει. Είναι σαφές ότι το πρωτόκολλο του Κιώτο θα έπρεπε να ε, εμπλέξει την ιδιωτική αγορά έτσι ώστε να πάρει μέρος στον καθορισμό ε, του κόστους των εκπομπών και να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο να είναι διαχειρίσιμο. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη απλά και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι όπως είπε και ο κύριος Μπελέτ στα πλαίσια της τροπολογίας του Της 8.21, ό,τι δηλαδή μπορούμε ε, εκ των προτέρων να ορίσουμε κάποια όρια για την χρήση της ενέργειας και ιδιαίτερα των ορυκτών καυσίμων, με τέτοιο τρόπο να περιορίσουμε την εκπομπή ε, καυσαερίων και ταυτόχρονα να καταστήσουμε με συγκεκριμένους κανονισμούς ε, πρακτική την ρύθμιση αυτή. Πολύ συχνά βέβαια οι υπορβολικές διακανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τα όρια των εκπομπών σαν παράδειγμα μπορεί να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Συνεπώς οφείλουμε να επανεξετάσουμε σε βάθος το πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Η επανεξέταση αυτή πρέπει να γίνει πριν το 2015 γιατί πολύ φοβάμαι ότι τα μέτρα τα οποία ακολουθήσαμε μέχρι τώρα δεν θα πετύχουν. <clears throat> Οφείλουμε με αρεαλιστικό τρόπο να θέσουμε το εξής ερώτημα αυτά τα οποία κάνουμε μέχρι τώρα πρέπει να τα συνεχίσουμε ή μήπως πρέπει να ακολουθήσουμε μία άλλη οδό. Ευχαριστώ κύριε Πρόντι. Τελευταίος ομιλητής, Πάσκα. Ďakujem Ευχαριστώ. Είμαι πισμένος πρέπει να πω για το γεγονός ότι θα πρέπει να τηρήσουμε αυτές τις ενδείξεις, ότι θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές ρήπων και να χρησιμοποιούμε περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να εξοικονομούμε ενέργεια. Από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι με αυστηρές τέτοιες προτάσεις και στόχους υπάρχει ο κίνδυνος στον οποίο μπορεί να εμπλακούμε η βιομηχανία να συρρυκνωθεί, να υπάρχει όλο και λιγότερος ανταγωνισμός, μικρότερη ανταγωνιστικότητα και να χάσουν τη θέση εργασίας τους οι εργαζόμενοι και να μετεγκατασταθούν σε άλλες περιοχές και περιφέρειες του κόσμου οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες. Γι' αυτό είμαι πεισμένος ότι η πολιτική μας στον ενεργειακό τομέα θα πρέπει να τροποποιηθεί, θα πρέπει να μεταβληθεί, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούμε ώστε λειτουργικά να μπορούμε να αντιδράσουμε αναλαμβάνοντας ε, πρωτοβουλίες αν κάτι είναι επιτυχές ή το αντίθετο αν κάτι πάει στραβά πάλι να μπορούμε να προσαρμοστούμε όπως χρειάζεται. Στόχος μας πρέπει πάντα να είναι να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Αυτό είναι ο στόχος μας. Και αν συμβαίνει αυτό τούτου λεχθέντος τότε μια ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να ακολουθηθεί που οικονομικά και χρηματοδοτικά μπορούμε πραγματικά να την ε, επομισθούμε, να την αντέξουμε και να την προαγάγουμε. Και θα πρέπει εδώ να δούμε και τους στόχους για το περιβάλλον. Σταθεροποίηση και σταθερότητα οικονομική και αυτό το οποίο είναι εφικτό οικονομικά να διαμορφώνει τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πάσκα την τελική σας φράση. Φτάσαμε στο τέλος των ομιλητών εξ του Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη ζητήσω να κάνει σχόλια όχι για όλες τις τροπολογίες, αλλά να μας δώσει κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία όπως ακούσατε και από τη συζήτησή μας μέχρι τώρα είναι, ε, θα έλεγα, κυρίαρχα Βλέπετε ποιο είναι το ύψος των ψηφιλοδοξιών μας, είδατε πού σταθήκαμε σε θέματα ανταγωνιστικότητας. Έχει τεθεί επανειλημμένα από τους ομιλητές και ε, ε, το, της τροπολογίας 821 του Μπελέτ για το τέλος αυτό. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ακούσαμε το όνομά του. Πρώτα θα μιλήσει η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ομιλώ εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης ε, Ενέργειας. Ε, είναι ένα κοινό εγχείρημα από πλευράς μας. Πρώτον το χαιρετίζουμε ότι υπήρξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και με τις 920 τροπολογίες που κατατέθηκαν πολλές πιστεύουμε ότι στοχεύουν στην ορθή κατεύθυνση. Φυσικά υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις όπως πάντα με ένα τέτοιο θέμα αλλά χαιρόμαστε ότι είναι δεδομένο το ενδιαφέρον και η προθυμία να συνεργαστείτε από ε, χρονικής είναι καλό γιατί τώρα βρισκόμαστε στη φάση προετοιμασίας αυτής της δέσμης μέτρων πράγμα που για την 22η Ιανουαρίου προβλέπεται ως ημερομηνία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσία στη συσκέψη έχουμε την φάση input, την φάση προτάσεων. Ενεργειακά για την πολιτική μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε απόλυτα με τους τρεις στόχους που αναφέρεται και τονίζεται. Ανταγωνιστικότητα και εδώ εννοούμε την ανταγωνιστικότητα για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις συνολικά ακόμα και μια πιο εντατική στην εκμετάλλευση της ενέργειας ε, βιομηχανία αλλά και με προσιτές τιμές. Αυτό είναι σημαντικό και για τη βιομηχανία και για τους χρήστες. Δεύτερον, είμαστε υπέρ της ασφάλειας του ανεφοδιασμού ενεργειακά και είμαστε υπέρ επίσης και της ε, ενεργειακής αποδοτικότητας. Και τώρα όσον αφορά τα μαθήματα, τα συμπεράσματα, φυσικά το ε, πακέτο 2030 δεν θα είναι το ίδιο με το πακέτο 2020. Διεξοδικά έχουμε ε, συζητήσει και έχουμε συλλέξει και πείρα με το πακέτο 2020 τις θετικές εμπειρίες και βιώματα σε σχέση με τους στόχους και υπάρχουν πολλές τέτοιες θετικές εμπειρίες αλλά και πράγματα από τα οποία μπορούμε να συναγάγουμε κάποια κριτικά συμπεράσματα. Αναφέρομαι αμέσω στο θέμα το οποίο εθίγει προηγούμενα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα ανανεώσιμα εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικά για μας και στο πλαίσιο των στόχων 2030. Είναι σαφές για μας ότι το κόστος της αποτελεσματικότητας πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη και μια αναγκαία αλλαγή, προσαρμογή νοοτροπίας πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, και μετά το 2030 σε σχέση με τις εργασίες μας για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ενέργειας και αυτό είναι πολύ σπουδαίο τμήμα των μέτρων 2030 αυτού του ορίζοντα Θα εξετάσουμε και άλλες επιπτώσεις άλλων μέτρων αλλά έχει υπόψη τον Ιούνιο 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται και με την ε, οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα πιθανότητα να δούμε αν χρειαζόμαστε συγκεκριμένο δεσμευτικό στόχο για το 2030 ή όχι. Ένα τελευταίο σημείο. Ενεργειακά κόστη και ενεργειακές τιμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πακέτο 2030 στις 22 Ιανουαρίου θα υποβάλει εξειδικευμένη καταλεπτός έκθεση όσον αφορά τις εξελίξεις και για τις τιμές και για την διαμόρφωση τιμών. Και αυτό ακόμα και για τα κόστη της ενεργοβόρου βιομηχανίας, της εντατικής στην εκμετάλλευση ενέργειας βιομηχανίας. Ε, και εδώ αρκετά πράγματα νομίζω ε, τίθενται σε ένα σωστό πλαίσιο ότι πρέπει τα κόστη να είναι προσιτά σε σχέση με τις, ε, τα, τα ορυκτά καύσιμα και οι τιμές αυτές των ορυκτών καυσίμων έχουν μεγάλη επιρροή σε όλα τα άλλα και αυτό θα το δούμε στα 28 κράτη-μέλη. Ποιος παράγοντας διαδραματίζει το μεγαλύτερο ρόλο και τι πολιτικά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι στα κράτη-μέλη μπορεί να επιτευχθεί. Ο κύριος Ρούγκας στη συνέχεια θα πει και άλλα πράγματα, ιδιαίτερα όσον αφορά άλλες πτυχές. Ευχαριστώ. I would like to ναι, θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω την προλαλή σας για τους ε, περιβαλλοντικούς στόχους. Καταρχάς, από την συζήτηση βλέπω ότι δεν έχουμε επιτυχημένη περιβαλλοντική πολιτική αυτή τη στιγμή. Όμως, ε, αντίθετα, τα στατιστικά στοιχεία μας δείχνουν ότι είναι πολύ επιτυχημένη η περιβαλλοντική πολιτική. Μέχρι από το 2008 μέχρι το 2012 είδαμε ότι έχουμε περίπου 8% μείωση σε σχέση με το 1990. Αλλά σήμερα είμαστε στο μείον 18% σε σχέση με το 1990. Και αυτή η μείωση κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έγινε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό όχι εξαιτία ε, τη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά ε, γιατί η ευρωπαϊκή οικονομία έχει γίνει πολύ πιο αποτελεσματική από ό,τι το 1990. Ε, αυτή λοιπόν είναι η επιτυχία που έχει ε, οδηγήσει στην ε, κατάρρευση των, ε, της τιμής του άνθρακα στο, στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργεια. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση δικαιωμάτων εκπομπής. Όταν υπάρχει υπερπροσφορά, χαμηλών, πέφτουν και οι τιμές. Και αυτό ακριβώ έχει γίνει και στην αγορά. Και φυσικά η χαμηλή αυτή τιμή δεν είναι κίνητρο σε καμία περίπτωση για καινοτομία, για ακριβές τεχνολογίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία. Τώρα, όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να πω ότι ορισμένες περιπτώσει έχουν δείξει ότι οι πολιτικοί που ακολουθούν τα κράτη-μέλη, και μιλώ για τα κράτη-μέλη διότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε θέσει έναν κοινό στόχο, η εφαρμογή όμω εξαρτάται από τα κράτη-μέλη και έχουμε 28 αυτή τη στιγμή διαφορετικέ πολιτικέ για την ανανεώσιμη ενέργεια. Ορισμένε από αυτέ είναι πολύ επιτυχημένε, όμω ε, έχουν παραλυφθεί ορισμένα στοιχεία, τα οποία ε, έχουν οδηγήσει σε αυτήν λοιπόν την ε, απόδοση κόστους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να διορθώσουμε. Και αυτό συμβαίνει και στη δική μου χώρα. Πώ δηλαδή να γίνει η πολιτική αυτή πιο αποδοτική. Και αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί και στο επόμενο πακέτο για το 2030. Πρέπει να υπάρχει αποδοτικότητα όσον αφορά την επίτευξη των ε, στόχων. Είναι όμω τελείω διαφορετικό να είσαι αποδοτικός χρησιμοποιώντας τα λιγότερα δυνατά μέσα για να επιτύχει του στόχου σου. Και αυτό προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά τους, ε, την ε, διαρροή άνθρακα και τους ε, στόχους και τους μηχανισμούς προσαρμογής δεν είναι λογικό να μεταφέρονται στόχοι, να μεταφέρονται δικαιώματα κομπών από το ένα κράτος στο άλλο. Αυτή δεν είναι σωστή περιβαλλοντική πολιτική. Πάντα θα έχουμε προκλήσεις όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Γιατί μπορούμε να μιλάμε για ε, ίσο και θυμητό ανταγωνισμό, είναι όμως πολύ δύσκολο αυτό να εφαρμοστεί στην πράξη. Υπάρχουν μικρέ διαφορέ. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορία Εκπομπών που έχουμε είναι κάτι που έχουμε δημιουργήσει για να αντιμετωπίσουμε την διαρροή του άνθρακα και αυτό έχει οδηγήσει στο να είναι η βιομηχανία μα εκτεθειμένη σε εξωτερικέ πιέσει, πιέσει από την παγκόσμια αγορά οι οποίοι δεν έχουν αυτό το σύστημα, έχουν ε, δωρεάν ε, κατανομή ε, των, και εκχώρηση των επιστοποιητικών αυτών. Η έκθεση λοιπόν και τα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή μας δείχνει ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε λόγο για διαρροή άνθρακα αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα ενώσο η τιμή του άνθρακα είναι πολύ χαμηλή. Τώρα, όσον αφορά το μηχανισμό προσαρμογής, συζητώντας το πρώτο πακέτο πολιτικής, υπάρχει στην αντίστοιχη οδηγία μία διάταξη που επιτρέπει τη δυνατότητα χρήσης παρόμοιων ε, μέσων έτσι ώστε να εξισορροπηθεί η αγορά. Όμως οι εμπειρίες που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικές με τη ρύθμιση μας έχουν δείξει ορισμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα έχουμε την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, όπου η ποιότητα των καυσίμων εξαρτάται από το σύνολο μια διαδικασία Και εδώ φαίνεται πόσο δύσκολο είναι να περάσει μια, ε, ένα τέτοιο μέτρο. Ο Καναδάς και πολλές άλλες χώρες αντιτίθενται σε αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα που πιστεύω ότι είναι και πολύ πιο ε, φανερό είναι η αεροπορία. Οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες έχουν συμπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα. Είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο φροντίζει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού και για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και για τις ε, διεθνείς. Και αυτό όμως είναι κάτι που ταυτόχρονα έχει οδηγήσει σε, ε, στην οργή των εταίρων μας, είτε της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε της Κίνας, είτε της Ινδίας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αυτή την ε, πρόταση στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά την επιτυχή συνεδρίαση του ΙΚΑΟ στο Μόντρεαλ. Υπέβαλε λοιπόν την πρόταση τροποποίησης του συστήματος και αυτό είναι μία ε, λύση του, του πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα. Ακόμα και εάν υπάρχει η νομική δυνατότητα, το ζητούμενο είναι η εφαρμογή. Πώς μπορούμε να φροντίσουμε τη σωστή εφαρμογή, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα προϊόν που έχει ε, δημιουργηθεί από ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμε και από ενέργεια που προέρχεται από ρηκτά καύσιμα. Αυτά είναι διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να επιληθούν. Και τέλο υπάρχει και η πολιτική διάσταση και προσωπικά πιστεύω ότι το, ότι η αντίδραση αυτή η έντονη αντίδραση της αεροπορίας είχε ως λόγο το ότι θεωρήθηκε ως το πρώτο στάδιο στο μηχανισμό προσαρμογής. Γι' αυτό λοιπόν πολεμούν με νύχια και με δόντια κάτι τέτοιο. Διότι φοβούνται το τι θα επακολουθήσει, τι θα προσπαθήσει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουν να δεχτούν. Ε, δείτε τι γίνεται, για παράδειγμα, με τις διεθνεί διαπραγματεύσεις για το περιβάλλον. Έχουμε τα κράτη-μέλη, τα οποία προσπαθούν να ρυθμίσουν τις εκπομπές αερίων στη δική τους επικράτεια. Και με το πρωτόκολλο του Κιώτο, και με την ε, διάσκεψη για το κλίμα και προσωπικά στην Βαρσοβία, στην ΕΚΟΠ δεν είδα κάποια ε, αλλαγή όσον αφορά την προσέγγιση. Είδα μόνο χώρες, είδα μόνο μέρη τα οποία διαπραγματεύονταν ως ε, κυρίαρχα κράτη. Αυτά λοιπόν από μένα. Εάν έχετε παραπάνω ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρούμ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευχαριστούμε επίσης και την κυρία Βέστερ, επίσης ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνεισήγητες θέλουν να ξαναπάρουν το λόγο για κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Κυρία Οκονή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύνολο των συναδέλφων για την ποιότητα της αναλύσεως τους και τον πολύ πλούσιο τρόπο με τον οποίο έχουν συνεισφέρει στη συζήτηση. Κάποια επιμέρους σημεία μετά από τις παρατηρήσεις τους. Για τον κύριο Αρολόταν λέτε ότι οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, αυτό το 20% δηλαδή, της στρατηγικής 2020 δεν είναι εντελώς σωστό. Οι στόχοι αυτοί προβλέπεται να τρέχουν μέχρι το 2020. Σήμερα βρισκόμαστε στο 2014 λέει η ομιλήτρια. Για το διοξίδιο του άνθρακα έχουμε ήδη φτάσει στο 17% για τις επόμενες γενιές. Στις ανανεώσιμες πηγές είμαστε στο 13% και μόνον στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας είμαστε σε ένα επίπεδο που δεν ξεπερνά το 10% αντί για 20%. Ακριβώς γιατί μέσα από την ενεργειακή αποδοτικότητα ο στόχος είναι ενδεικτικός, όχι ε, υποχρεωτικός. Γι' αυτό λοιπόν όταν έχουμε στόχους εσμευτικούς έχουμε αποτελέσματα θετικά. Και δεν μπορώ να δεχθώ ότι βρίσκεται σε αντιπαράθεση ένα κάποιο όραμα περιβαλλοντικό με την αποδοτικότητα. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωνέας ενέργειας στον κόσμο και από το 2011 έχουμε εισάγει το 50% και άνω της ενέργειάς μας. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο πράγμα, ένα κόστος για τις επιχειρήσεις μας και τελικά για τους πολίτες μας και θα πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν. Υποχρεωτικά διαπιστώνουμε σήμερα ότι αυτές οι διαφορετικές πολιτικές που συνδέονται με την καταπολέμηση των συνεπειών της υπερθέρμανσης και της μείωσης, της προσπάθειας της μείωσης ε, του διοξιδίου του άνθρακα, όπως επίσης και της αναζήτησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, έχουν δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες απασχόλησης, ενώ σε άλλους τομείς βλέπουμε ότι δυστυχώς έχουμε χάσει και σημεία ανάπτυξης και θέσεις απασχόλησης πάρα πολλές. Θυμίζω ότι μέχρι την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για το 20 θα δημιουργηθούν 20 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, οι στόχοι λεγόμενοι τρεις φορές το 20 υπογραμμίσατε όλοι επανειλημμένα τη σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας. Εδώ θα πρέπει να περάσουμε από στόχους όμως για να το πετύχουμε δεσμευτικούς. Για την κυρία Φιώνα Χολ, πράγματι αυτό που είπατε ε, είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής, συμφωνώ μαζί σας, πράγματι μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση, και ακολουθώντας τον δρόμο της αποδοτικότητας θα κερδίσουμε ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις μας, για την κυρία Χιόξκοκ που λέει ότι η 2.90 είναι τροπολογία του ΕΛΚ δηλαδή συντηρητική διότι απαιτεί μια στάση αναμονής για τις αποφάσεις του COP21. Εδώ θέλω να πω που θα οργανωθεί στο Παρίσι ότι η τροπολογία αυτή αντιπροσωπεύει κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και σε καμία περίπτωση δεν είναι η επίσημη γραμμή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είμαι πεπισμένη όπως και εσείς ότι απαιτούνται στόχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να περιμένουμε τον υπόλοιπο κόσμο αλλά για να αποδείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σημαντική είναι η επίτευξη των στόχων αυτών και για την ανταγωνιστικότητα. Και συμφωνώ με την τροπολογία Μπελέτ που ζητά να υπάρξει μια φορολογική ρύθμιση στα σύνορα, διότι τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με προέλευση άλλες χώρες εκτός της Ένωσης και που δεν υπόκεινται στους ιδίους περιβαλλοντικούς όρους θα πρέπει προφανώς να υποβάλλονται σε ένα συγκεκριμένο φόρο και εκεί θα λύσουμε το θέμα του αθέτημι του ανταγωνισμού. Είναι απαράδεκτο οι επιχειρήσεις μας να υποβάλλονται σε φορολογικές επιβαρύνσεις για να πετύχουμε τη μείωση των εκπομπών και από την άλλη να δεχόμαστε προϊόντα τα οποία παράγονται με συνθήκες εντελώς ευνοϊκές να εισέρχονται χωρίς φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν πάση περιπτώσει ε, συμφωνώ με την τροπολογία του κυρίου Μπελέτ που έχω συνυπογράψει. Να πω εδώ στον κύριο Σιμάνσκι, είπατε ότι απαιτείται περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση της εξάρτησής μας. Ναι, Ιδιαίτερα στον τομέα των ορυκτών καυσίμων αυτό είναι απαραίτητο. Επαναλαμβάνω, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι θα πλήρως εξαρτημένη από τις εισαγωγές ε, ορυκτών ε, καυσίμων και αυτό ε, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι περισσότερο να πω, δεν είμαι βέβαιη ότι κάτι δεν ξέχασα, αλλά εν πάση περιπτώσει σταματώ εδώ. Ευχαριστώ την κυρία Οκονή θα δώσω το λόγο στον κύριο Σουμάνσκι. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Για αυτή τη συζήτηση ευχαριστώ. Πιστεύω ότι μπορούμε όλα να τα εντάξουμε σε ένα κοινό παρονομαστή, την αηφορία, την ανάπτυξη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συνδυάσουμε και να τα συνδέσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι κέρια σημασία θέματα. Είναι και θέματα στρατηγικής. Πρέπει να εξευρεθεί μια τέτοια μέθοδος ώστε όλοι αυτοί οι στόχοι να μπορέσουν να ενταχθούν σε ένα κοινό πλαίσιο. Και αυτό είναι, αυτή είναι η στόχη που σε αυτή την πολιτική συμφωνία αναπαριθμούνται, αναφέρονται δεν είναι θέμα πρόκλησης εδώ αν επαναλάβουμε τις θέσεις των κρατών μελών σε κάποιους στόχους αηφορία, ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια ανεφοδιασμού, ενεργειακή ασφάλεια. Όλα αυτά θα πρέπει σε αυτό το πακέτο να υλοποιηθούν. Δεν είναι απλά και μόνο το θέμα της ασφάλειας ε, ή στον ανεφοδιασμό ή κάποιων ξεχωριστών θεμάτων. Όχι. Πρόκειται για κάτι πολύ παραπάνω. Πρέπει να καταδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικά δυνατόν και είναι με αηφορία δυνατόν να λειτουργήσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η ανταγωνιστικότητα και η ενεργειακή ασφάλεια ανεφοδιασμού δεν πρέπει να αμεληθούν, δεν πρέπει να αγνοηθούν. Στατιστικά στοιχεία αναφέρονται. Αναφέρονται θέματα για την ίδια την βιομηχανική παραγωγή. Δεν είναι θετικό παράδειγμα κάτι τέτοιο για ε, όλο τον κόσμο. Πολλά κράτη δεν πιστεύουν ότι η Ευρώπη πραγματικά μπορεί να είναι πρότυπο. Γι' αυτό τον λόγο στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία και αλλού σήμερα έχουμε μία επανάληψη και επιστροφή αυτής της εξέλιξης και πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε με αηφορία να συνδυάσουμε αυτούς τους στόχους. Την ασφάλεια του ανεφοδιασμού, την ζήτηση, την κάλυψη των αναγκών και την ανταγωνιστικότητα και την αηφορία. Σήμερα ε, δεν έχει γίνει ακόμα κάτι τέτοιο. Κάνουμε λόγο για αυτούς τους στόχους ε, και πρέπει να μπορέσουμε να τους συνδυάσουμε. Και δυστυχώς η μονομέρεια, ο μονομερής χαρακτήρας από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ε, κλιματολογικά θέματα δεν θα μπορέσει να κερδίσει κανέναν και να τον ε, ε, σε εισαγωγικά προσιλητήσει. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι αυτό το οποίο αφορά τη βιομηχανία τους διάφορους ε, τομείς της βιομηχανίας. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, ιδιαίτερα για την ενεργοβόρα βιομηχανία, την σε ένταση ε, χρήση ενέργειας ε, από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες. Τώρα, σε σχέση με τέλη, με ειδικά τέλη, αυτό μια ολόκληρη, ένα μια ολόκληρη σειρά διαμαρτυριών μπορεί να προκαλέσει και στο επίπεδο του ΠΟΕ, Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά και εκτός αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προανέφερε ότι στον τομέα των εναέριων μεταφορών υπήρξαν αυτές οι προσπάθειες για αυτά, την εισαγωγή αυτών των τελών και απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν δείχνουν καμία προθυμία και δεν είναι καθόλου έτοιμες και πρόθυμες αυτές οι χώρες να συνεργαστούν. Και δεν είναι δυνατόν να είμαστε με μονομένη νησίδα, απομονωμένη νησίδα εμείς ε, σε παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά ξεχωριστή πρωτοβουλία ή δράση που θα αναπτύσσαμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι η Ήπειρός μας, η Ευρώπη, πάντα βασιζόταν στο εμπόριο. Και σήμερα με βάση μια ανοιχτή οικονομία, παγκόσμια οικονομία, όπως δρούμε, επειδή ενεργά συμμετέχουμε στο παγκόσμιο εμπόριο, πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη συνιστόσα. Αυτό που περιπλέκει ιδιαίτερα τα πράγματα είναι τα θέματα των ενεργειακών τιμών η τιμολόγηση, ας το πω έτσι, των ενεργειακών προϊόντων. Πολλοί βιομηχανικοί τομείς, όχι μόνο οι ενεργοβόροι τομείς, αλλά και αλλού βλέπουμε ότι η υλοποίηση αυτών των στόχων ταυτόχρονα δεν ε, έχει οδηγήσει στα ε, πιο θετικά αποτελέσματα. Έχουν διαφορετικό δυναμικό τα κράτη-μέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα στην χρήση ενέργειας. Σε κάποιες ε, χώρες μας έχουμε μεγάλο δυναμικό και μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το δυναμικό όμως είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο θα διεξαχθεί ένα σεμινάριο τον Ιανουάριο προτού ψηφίσουμε προς έγκριση ώστε εκπρόσωποι των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων θα προσέλθουν εδώ στις Βρυξέλλες και θα μας αναφέρουν ποια είναι τα βιώματά τους, η πείρα που έχουν συλλέξει και το τι συμβαίνει από πλευράς τους δεν θέλουμε να έχουμε μια μετοπική αντιπαράθεση. Όχι, το αντίθετο. Θέλουμε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Συμβιβασμούς που θα μας επιτρέψουν στην Ευρωβουλή να καταλήξουμε σε 75% συνένεση υπέρ του ανοίγματο ε, της πολιτικής που θα υιοθετηθεί προς αυτούς τους στόχους, ώστε να δείξουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη, η αηφορία και η ασφάλεια ανεφοδιασμού ως οι τρεις αυτοί στόχοι μπορούν να συνδυαστούν και να ε, ολοκληρωθούν. Έχουμε ένα πολύ καλό δυναμικό και πολλές δυνατότητες. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σουμάνσκι, ευχαριστώ επίσης και την κυρία Οκονή για τις παρουσιάσεις τους, ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμίζω ότι η επόμενη συνάντηση κοινή των επιτροπών μας ε, για να περάσουμε στην ψηφοφορία την 9η Ιανουαρίου. Προβλέπονται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια ε, στις 6 Φεβρουαρίου. Σας ζητώ από όλους να συνεχίσετε τις προσπάθειες ε, για να καταλήξετε σε ικανοποιητικές ε, συμβιβαστικές τροπολογίες λόγω του υψηλού αριθμού των κατατεθειμένων τροπολογιών μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου για να μπορέσουμε έτσι να σεβαστούμε ε, τις διαδικασίες και να ψηφίσουμε με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Σας ευχαριστώ όλους όσους πήρατε μέρος. Τερματίζονται οι εργασίες μας, θα τα ξαναπούμε.